κοντά ασύμβατα, με το έργο του Ευρωβουλευτή. το διορθωτικό ε, σύμφωνα με το άρθρο 216 του κανονισμού η Επιτροπή Μεταφορών μετέφερε το παρακάτω διορθωτικό σχετικά με ένα κείμενο που ανέκρινε το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα διορθωτικό στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 27η Σεπτεμβρίου 2011 που αφορά την οδική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την περίοδο 2011-2020. Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό ε, ε θεωρείται πως εγκρίνεται εκτός εάν εντός ε, των προσεχών 48 ερών μια πολιτική ομάδα ή 40 βουλευτές τουλάχιστον ζητήσουν να ψηφιστεί. Σήμερα λοιπόν δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Δηλώνω πως ε, το διορθωτικό κατατέθηκε και έχει 48 ώρες ε, για να ζητήσετε ενδεχομένως την ψήφιση του και μπορείτε να το βρείτε στην ε, ιστοσελίδα Seons on Direct. Η κυρία Ροτ Μπέρεντ επιθυμεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριος Λάιτφριντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι κατάλληλη χρονική στιγμή ίσως, αλλά σκέφτηκα... Ε, δεν μπορούσα να βρω κάποια πιο κατάλληλη στιγμή ο συνάδελφος Φαχών μου ε, επεσήμανε και ελπίζω να μην υπάρχει κάποια άλλη αιτία ότι τα ονόματά μας δεν φαίνονται πλέον και δεν ξέρω αν είναι αυτή η θέση μου επειδή ζητήσατε την... είπατε να πάρει το λόγο η κυρία Ροτ Μπέρεντ δεν ξέρω μήπως κάτι έχει γίνει λάθος με τα έντρανα και την ονομασία των εντράνων Ίσως θα μπορούσατε να φροντίσετε να το ελέγξουν οι κατάλληλες υπηρεσίες Μάλιστα θα ελέγξουμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση και την πληροφορία που μου δώσατε. Έλαβα από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, και από την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς ε, τήσεις για διορισμούς στις επιτροπές και τις κοινωνικές ελπισοπίες. Ο κατάλογος των